για μια συγγνώμη, διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη. Θα σας δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πρόταση για μια νέα διαστημική στρατηγική και τους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές για την συνεισφορά τους σε αυτό το σημαντικό θέμα έχουμε τεράστιες δυνατότητες που πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε. Το διάστημα πλέον δεν είναι κατομακρινό, επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα δεδομένα του Κοπέρνικου χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην θύελα η οποία πλήττει την Καραϊβική και την Φλόριδα. Υπάρχουν όμως ε, και άλλοι τομείς εφαρμογής, ε, η κλιματική αλλαγή, η παρακολούθηση των εκπομπών, διοξιδίου του άνθρακα, μεθανίου, ε, της αλληλείας, ε, μεγάλων ε, οικοδομικών έργων όπως η γέφυρα μεταξύ Δανίας και Σουηδίας που χτίστηκε με δεδομένα από ευρωπαϊκούς δορυφόρους για να καταφέρουν να συναντηθούν από τις δύο άκρες. Επίσης τα σύγχρονα συστήματα, τα συστήματα πλοήγησης τα οποία εξαρτώνται αυτή τη στιγμή ακόμα από τη ΣΥΠΑ. Αλλά και η συνδεσιμότητα απομακρυσμένων ε, περιοχών με γρήγορο ίντερνετ μέχρι την αντιμετώπιση της ε, προσφυγικής ε, κρίσης. Όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν με στήριξη από το διάστημα. Για όλα αυτά χρειάζεται μια έξυπνη στρατηγική για το ποιο θα επενδύσει τι σε ποιου τομεί. Οι προτάσει Κομισιόν είναι μπροστά σα. Έχουμε συζητήσει την έκθεση και επεκτείνει τις προτάσεις. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη χρήση των δεδομένων από το διάστημα και πρέπει να το προωθήσουμε αυτό και στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. Πρέπει να βελτιωθεί και η επικοινωνία και η εκπαίδευση επίσης γιατί δεν είναι γνωστό ακόμα για πολλούς το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα και τι μας προσφέρουν όλα αυτά. Τα ήδη υφιστάμενα έργα πρέπει να συνεχίσουν και να επεκταθούν. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του Γαλιλαίου, του Έγνος και του Κοπέρνικου. Ε, όχι μόνο στον ε, τομέα των κοινωνικών αλλά και στον οικονομικό. Στη διαχείριση της, κληρονομ... της κυκλοφορίας ε, των υδάτων ε, στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών από νεοφυείς επιχειρήσεις ανοίγεται ένα πεδίο δόξης λαμπρών για την χρήση αυτών των δεδομένων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να στηριχθούν και, εάν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να νομοθετήσουμε. Επίσης, θα πρέπει να κινητοποιηθούν και οι τοπικοί φορείς ε, για να εκμεταλλευτούν αυτά τα δεδομένα, παραδείγματο χάρη στην πολεοδομία ή στην προστασία από καταστροφές, στην πολιτική προστασία. Και όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα συνεχίσουμε να είμαστε παγκοσμίω ανταγωνιστικοί και βεβαίω να υπάρξει και η κατάλληλη οικονομική πλαισίωση των προγραμμάτων μας. Χρειαζόμαστε στο και στο μέλλον έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για διαστημική πολιτική, ο οποίος δεν θα μειωθεί. Αντιθέτως, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής οι δορυφόροι και βλέπουμε πως είναι σαφώς μεγαλύτερες οι επενδύσεις των ΙΠΑ εδώ πέρα. Βεβαίω, σημασία έχει η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, της ΕΖΑ και των ε, κρατών μελών. Όπως παραδείγματο χάρη μέσω του προγράμματος ορίζοντας του ερευνητικού προγράμματος. Και ε, βεβαίω ε, θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για το πρόγραμμα άμυνα και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν αύξηση του αριθμού μικρών και μεγάλων δορυφόρων, κάτι το οποίο μπορεί να σημάνει και κίνδυνο από κυβερνοεπιθέσεις. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να κινητοποιηθούμε. Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Ένωσης και της ΕΖΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους στόχους αλλά και μια στρατηγική επικοινωνία. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε το Catch the Eye με τον κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ υποδέχομαι θετικά την πρόταση της ε, Επιτροπής που θέλει να λάβει δράση σε αυτή την διαστημική στρατηγική και από την πράγα έτσι το βλέπουμε η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε συνδέεται φυσικά και με το διάστημα και μάλιστα πολύ καλά τα είπε η συγγήτρια έχουμε εδώ να αναπτύξουμε πάρα πολλά στοιχεία όμως εγώ θα ήθελα να μιλήσω κυρίως για τις startups, για τις νοσίστατες επιχειρήσεις, αλλά όχι και μόνο. Θέλω να μιλήσω και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, και για τους δικαιούχους των προγραμμάτων. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που τόνισε και το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκηση και των περιφερειών ε, για να μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις τεχνολογίες για την ανάπτυξή τους. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καινοτόμος αυτή η προσέγγιση και θέλω να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Ευχαριστώ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 η έκθεση που θα υιοθετήσουμε συνεισφέρει στη χάραξη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη. Είναι στρατηγικό τομέα ε, που δυστυχώ όμω αγνοείται από την κοινή γνώμη. Ο διαστημικό τομέα στην πραγματικότητα δεν αποτελεί κόστο για του πολίτε, αλλά επένδυση. Τα διαστημικά προγράμματα ε, και οι υπηρεσίε αποτελούν ε, τροφοδότηση για πάρα πολλού τομεί όπω η υγεία, οι μεταφορέ, το περιβάλλον, η ψηφική αγορά, η επικοινωνία και πάρα πολλά άλλα. Για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει. το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη πρικοδότηση για το διαστημικό τομέα. Πρέπει να συνεχιστούν τα προγράμματα και να σκεφτούμε για το πώ θα εξελιχθούν ο Κοπέρνικο και ο Γαλιλαίος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα για τι επενδύσεις στον τομέα. Παρ' όλα αυτά δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον ευάλωτο χαρακτήρα των διαστημικών υποδομών, οι οποίε ε, μπορεί μπορεί να υποστούν επιθέσεις ή παρεμβολές. Πρέπει να εγγυηθούμε την ύπαρξη των υποδομών αυτών και να αναπτύξουμε αρθρητικές τεχνολογίες. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το διάστημα δεν δύναται σήμερα να αντιμετωπιστεί απλώς σαν μια ακόμη αγορά για τους ιδιώτες επενδυτές. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανεύθυνο οι αποφάσει που αφορούν το διάστημα επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των χωρών αλλά ενδέχεται να έχουν και μακροπρόθεσμε συνέπειε στο φυσικό περιβάλλον. δεν δύναται λοιπόν να γίνει το διάστημα μια αγορά όπω όλε οι άλλε. διαστημικέ τεχνολογίε έχουν προστιθέμενη αξία για πολλού τομεί όπω οι τηλεπικοινωνίε και οι μεταφορέ. έτσι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζει το διάστημα με τι ίδιε ιδεολειψίε που αντιμετωπίζει και του υπόλοιπου τομεί κοινή δράση πρώτα απ' όλα η πολιτική του διαστήματο συνεπάγεται έρευνα δηλαδή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. τέλος η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να συνεργαστεί στον τομέα του διαστήματο, όχι μόνο με τι Ηνωμένε Πολιτείε και την ιαπωνία αλλά και με άλλε διαστημικές δυνάμει όπω η κίνα η ινδία και η ρωσία προκειμένου να έχουν ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα στη διαστημική τεχνολογία εχμής και επίση θα πρέπει όλα αυτά να τεθούν στην υπηρεσία τη ανθρωπότητα. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 1967 ο ΟΗΕ κατέληξε στην ε, Διεθνή Σύμβαση του Διαστήματος. Εν τω μεταξύ βεβαίως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και στηρίζουμε πλήρως την έκθεση και τα όσα αναφέρει τον Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο τα προγράμματα αυτά και πρέπει να αφιερώσουμε και τους κατάλληλους πόρους γιατί η δορυφορική επιτήρηση μας βοηθάει στην καθημερινή μας ζωή. Εγώ όμως θα ήθελα να πάω ένα βήμα παραπέρα. Θα ήθελα να σας πω πως ε, οι ΙΠΑ δήλωσαν ότι θα ενθαρρύνουν ε, τον ιδιωτικό τομέα να αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώματα σε ορισμένα σημεία του φεγγαριού. Ε, ανάλογες φιλοδοξίες για την σελήνη έχει και η Κίνα. Γι' αυτό είχα θέσει ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Πώς θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σελήνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το διάστημα έπαψε πλέον να αποτελεί ε, ένα, μια άγνωστη περιοχή η οποία δημιουργεί φόβο και δέος στον άνθρωπο. έχει πλέον προσεγγιστεί έχει ερευνηθεί και χρησιμοποιείται προκειμένου να παρέξει πλεονεκτήματα στην κοινωνία. το διάστημα επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή μας δίνει πρόσβαση σε επιτεύγματα της τεχνολογίας μας δίνει πολλές πληροφορίες με τους δορυφόρους που υπάρχουν επάνω σε αυτό και γενικά μπορεί αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα να δημιουργήσει και θέσεις εργασία. πάνω απ' όλα όμω επηρεάζει και την πολιτική και γι' αυτό ακριβώ το λόγο πρέπει να γίνει μια προσεκτική στρατηγική σχεδίαση για την επικοδομητική χρησιμοποίηση του διαστήματο από την ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με άλλε χώρε οι οποίε έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τεχνολογία να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα αυτού του σχεδιασμού και γενικώ να δώσουν την διάσταση της επιτυχίας και της προοπτικής στις σχέσεις του διαστήματος με τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ε, Ολοκληρώνεται εδώ το Κατσιλιά. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την ε, εξαιρετική εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση. Τον περασμένο Οκτώβριο η Κομισιόν υιοθέτησε τη διαστική στρατηγική για την Ευρώπη. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη σε αυτό το τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στείλαμε ένα σαφέ μήνυμα ότι το διάστημα είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν και η στρατηγική αποτελεί σαφή φιλοδοξία να καταστήσουμε την Ευρώπη ένα πρωταγωνιστή στο διάστημα. Χαιρόμαστε που υποστηρίζει η έκθεση αυτό το επίπεδο φιλοδοξία και μάλιστα πηγαίνει και μακρύτερα. Η έκθεση υιοθετεί πλήρω ε, την άποψη Τη της Κομισιόν και θέτει επιτόπου συγκεκριμένες προτάσεις, επιτάπητο συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με τις ε, τέσσερους στόχους, πώς ε, θα βελτιώσουμε τα ωφέλη της διαστημικής στρατηγικής για την οικονομία και για τους πολίτες, πώς να προωθήσουμε έναν ανταγωνιστικό διαστημικό τομέα, ε, να διασφαλίσουμε αυτόνομη πρόσβαση της Ευρώπη στο διάστημα και να ενδυναμώσουμε την Ευρώπη ως παγκόσμιο παίκτη. Η εφαρμογή της στρατηγικής ήδη ξεκίνησε και ήδη φέρει ωφέλη. Όλα τα διαστημικά μας προγράμματα είναι λειτουργικά. Το τελευταίος δορυφόρος ε, του Κοπερνικού έχει εκτοξευτεί και τα στοιχεία χρησιμοποιούνται ήδη ε, σε διάφορες επιχειρήσεις διάσωσης. Οι ε, υπηρεσίες του ε, Γαλιλαίος ε, ξεκίνησαν ε, τον περασμένο Δεκέμβριο. Ήδη, ήδη έχουμε 13 μοντέλα σε smartphones που λειτουργούν με τα σήματα του Γαλιλαίου. Το έγνος έχει δείξει την προσθεμένη αξία του. Σήμερα έχουν αναπτυχθεί project σε 182 αεροδρόμια το ε, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ε, την ανείχνευση έχει λειτουργήσει και ουσιαστικά δημιουργεί μια κατάσταση λιγότερης εξάρτησης. Αυτά είναι καλά, αλλά δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Φέτος και τα επόμενα δύο έτη θα είναι ζωτική σημασία. Θέλουμε να υιοθετήσουμε δράσεις στη διαστημική στρατηγική και θέλουμε να έχουμε την ίδια ολοκληρωμένη διαδικασία που ακολουθήσαμε την προετοιμασία της μελέτης. Οι προτεραιότητες μας είναι καταρχήν ε, για την δίσδυση στην αγορά. Ήδη διάφοροι πρωταγωνιστές ε, χρησιμοποιούν ε, τις εφαρμογές του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου. Δεύτερον, θέλουμε να προωθήσουμε ε, τις νοσίστες της επιχειρήσεις με συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε πιο αποτελεσματικές δαπάνες για το διάστημα και να αναπτύξουμε και τις ΔΙΤ. Τρίτον, πρέπει να προετοιμάσουμε την συνεχή εξέλιξη του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου. Αυτό θα ξεκινήσει με μια αξιολόγηση του τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τέταρτον, οι συνέργειε μεταξύ τη διάσταση ασφάλεια και άμυνα θα πρέπει να ενισχυθούν. Παραδείγματο χάρη να υπάρχει και συνδέσμο με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα και η μεταρρύθμιση του SSD θα λάβει υπόψη αυτή τη διάσταση. Επίσης, η αυτόνομη πρόσβαση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και τέλος να μην ξεχνάμε τις ε, πτυχές διακυβέρνησης και ότι πρέπει να συνεργαστούν ε, όλοι οι φορείς και πρέπει να συνεργαστούμε ιδίως με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Αυτές οι προτεραιότητες θα αντικατοπτριστούν τα επόμενα χρόνια σε νομοθετικές προτάσεις. Όμω ε, πρέπει να δούμε και το θέμα του προπολογισμού. Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και μελλοντικέ προκλήσεις. Όπως περιγράφει η έκθεση, ε, οι εφαρμογές οι διαστημικές εξυπηρετούν τους πολίτες και το διάστημα δεν αποτελεί κόστος αλλά επένδυση. Α εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα υποφεληθεί πραγματικά από τις επενδύσεις αυτές. Ας εργαστούμε για να πετύχουμε μια ισχυρή Ευρώπη στο διάστημα και ε, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα τομέα όπου δεν μπορεί ένα μόνο ευρωπαϊκό φορέα να πετύχει, αλλά χρειάζεται κοινή δράση.